Πάμε τώρα στις ε, επεξηγήσεις ε, ψήφου. Για την έκθεση Ταβάρης, ο κύριος ε, Κλέης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταψήφισα την έκθεση Ταβάρας για την εισαγωγή Ενό ε, νέου ευρωπαϊκού προγράμματο επανεγκατάσταση. Είναι ένα νέο βήμα σε μια νέα ε, ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Δεν χρειάζεται να είναι μάντη για να ξέρει ότι αυτό θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των υποψηφίων των ζητούνων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η εισαγωγή τέτοιου Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εμπανεγκατάσταση θα οδηγήσει, λέει η έκθεση, στο να είναι λιγότερο ελκυστική η Ευρώπη για τους παράνομους μετανάστες. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι σωστό. Είναι επιχείρημα που χρησιμοποιείται πάντα όταν εξετάζουμε θέματα ε, ασύλου, αλλά είναι σαν να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Στο Βέλιο ότι γίνονται εδώ, ζητάνε άσυλο, δεν τους δέχονται, και παρόλα αυτά παραμένουν. Λοιπόν, αυτό το ευρωπαϊκό πρόβλημα δεν, πρόγραμμα δεν είναι λύση. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτοβα. Ρόιτοβα. Κυρία Πρόεδρε, αυτή η οδηγία την οποία εγκρίναμε ε, προσφέρει εν πάση περιπτώσει νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής ε, απόδοσης σε διάφορα κτίρια. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στα παλιά κτίρια. Εδώ λοιπόν είναι απαραίτητο να βρούμε μια λύση έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων γιατί βεβαίως μέχρι το 2014 μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση. Πάμε τώρα ε, στην ε, επόμενη έκθεση και έχω πάλι την κυρία Ρόιτοβο για την έκθεση Κοέλιο. Κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ζήτησα το λόγο για το θέμα του Ταμείου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ είμαι σαφώς υπέρ της ε, αποδοχής ε, των νόμιμων μεταναστών και πρέπει να βελτιώσουμε τα σχετικά μέτρα ακόμα και μέσα στις χώρες Schengen. Ε, Σήμερα αποφασίσαμε για νέα μέτρα για την δεύτερη εκδοχή του συστήματος Schengen το οποίο πρέπει να βελτιώσει τη ζωή όλων όσοι ζουν μέσα στην περιοχή αυτή. Ε, βεβαίως ε, η πρακτική της ε, γερμανικής και της αυστριακής αστυνομίας δημιουργεί προβλήματα γιατί πάρα πολλοί Τσέχοι υφίστανται περί τους ελέγχους. Πριν από δύο χρόνια εγώ επισήμανα στην Κομισιόν αυτό το ατυχές γεγονός και μέχρι τώρα δεν έχει εξευρεθεί λύση. Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των υφιστάμων κανόνων και παραβιάζει την ελεύθερη μετακίνηση των ε, τσέχων επιχειρηματιών. Όμως η ελεύθερη μετακίνηση είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Κύριε Μαστέλα, κύριε Πρόεδρε, μια μεταναστευτική πολιτική που θέλει να είναι η ρεαλιστική πρέπει να προβλέπει ε, και τη δυνατότητα ασύλου και ρεαλιστικά προγράμματα. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η επανένταξη, η ένταξη δεν είναι ε, μόνο ανθρωπιστικό θέμα, αλλά είναι και οικονομικό, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις ε, χώρες εκείνες που μπορούν να δεχθούν πίσω τους μετανάστες. Και θέλω να πω ότι μία γραμμή στον προπολογισμό δεν αρκεί Γι' αυτό λοιπόν τα κράτη-μέλη πρέπει να προβλέψουν μηχανισμούς απαραίτητους για να ενθαρρύνουν και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε ο στόχος τελικά είναι να προαχθεί αυτή η ε, λήψη μέτρων. Είναι απαραίτητο να προβλέπονται και ad hoc ε, κονδύλια εμείς λοιπόν προτείνουμε να υπάρχει ουσιαστική δέσμευση όλων των άμεσα εμπλεκόμενων έτσι ώστε να υπάρχουν και οι σωστοί καταβλισμοί, οι δυνατότητες να μάθει κανείς τη γλώσσα και οι θέσει εργασίας. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να υπάρχει μια ε, ε, ε, ενσωμάτωση των μεταναστών χωρίς προβλήματα. Ο κύριος Κέις. Φαίνεται ότι έχει φύγει από την αίθουσα. Προχωρούμε στην έκθεση Λούλινγκ. Η κυρία Ροϊτόβα πάλι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι διότι η έκθεση για την ισότητα των φύλων έτυχε πολύ ευρεία στήριξη σήμερα. Όντως είναι ευθύνη των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι οι αυτοαπασχολούμενες ε, γυναίκες έχουν τη σωστή ε, προστασία και κοινωνική ασφάλιση. Βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να σέβονται ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν σημαίνει ότι παραβαίνουμε την αρχή της επικουρικότητας. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουν τα εθνικά κοινοβούλια αυτή την επιλογή και περιμένω να δω κατά πόσο θα αξιοποιηθεί αυτή η επιλογή ή θα συνεχίσει αυτή η ατέρμονη κριτική εναντίον της. Κύριε Τρικένα, κοίταξε, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι γυναίκες παίρνουν 17,4% λιγότερο ε, ρομίστιο από ότι οι άντρες και η διαφορά αυτή μειώθηκε τα περασμένα χρόνια. Σε άλλες χώρες όμως μεγάλωσε. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση να υπάρξουν τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις για τη διαφορά, τη μισθολογική μεταξύ ανδρών και γυναικών και για τις εκκρίσεις κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Πολύ ωραία για την ίδια έκθεση κυρία Ροϊτόβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλώντας για αυτό το θέμα, πολλοί συνάδελφοι είχαν υποβάλει άλλες προτάσεις προς εξέταση από την Ολομέλεια. Για παράδειγμα, να διευρυνθεί η πρόβλεψη και σε άλλους τομείς. Μιλούμε για τεχνικούς ορισμούς εδώ και χρειαζόμασταν την ε, βοήθεια, την τεχνική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και δεν ψήφισα υπέρ και θέλω να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παρουσιάσει πιο συγκεκριμένε και έγκυρες προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με την έκθεση αυτή θα ήθελα να πω ότι δεν μπόρεσα να ψηφίσω υπέρ των προτάσεων αυτών γιατί πιστεύω ότι συνηγορούν στον προστατευτισμό. Ευχαριστώ κύριο Σκροπότσκι. Για την έκθεση Άλβαρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ υπερψήφισα αυτή την πρωτοβουλία, διότι θεωρώ ότι έτσι δίνουμε ευκαιρία να αναπτυχθούν περισσότερο συγκεκριμένε περιφέρειες τη Ευρώπη. Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης ε, αντιμετωπίζουν οικονομικέ δυσκολίε τι οποίε πρέπει να γνωρίζουμε και πρέπει να κατανοούμε. Είναι και αυτέ μέρο τη Ευρώπη και του αξίζουν ίσες ευκαιρίε, Οι ευκαιρίε που επιφυλάσσουμε στι άλλε περιφέρειε. Συμφωνώ λοιπόν με αυτά τα προγράμματα τα αναπτυξιακά ε, και για την Γεωργία και για την Αλία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιντρία για την έκθεση Άλβες πάλι. Για την έκθεση Άλβες επαναλαμβάνω. Γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, για αυτό το θέμα δεν θέλετε να μιλήσετε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκφράζω την ανησυχία μου για την κατάσταση των παραγωγών μπανάνας στις Κανάριες νήσους σε σχέση με τους παραγωγούς του ίδιου προϊόντος στη Μαρτινίκα και του Γουαδελούπη κατάσταση έχει επιδεινωθεί ειδικότερα μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ε, ΠΟΕ με τις ε, λατινοαμερικανικές χώρες για εισαγωγές από εκείνες τις χώρες. Το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταρρυθμίσε ε, την κοινή οργάνωση αγοράς για τις μπανάνες και έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο δεσμεύει 208 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών μπανάνας στις Κανάριες νήσους, στις Αζόρες, στη μαντέρα, μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να συμφωνούμε με αυτή τη στήριξη. Ωστόσο δεν είναι αρκετή. Καλό λοιπόν τα αρμόδια θεσμικά όργανα να θετήσουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ένας τόσο παραδοσιακός οικονομικός κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, διακινδυνεύσει το μέλλον του ε, λόγω των ε, συμφωνιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στηρίζω την έκθεση αυτή γιατί λύνει το θέμα της διαφοροποίησης της ποικιλότητας στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης. Ωστόσο, εκφράστηκαν ανησυχίε για την επανέναρξη των συνομιλιών με τι χώρε Μερκοσούρ και συμφωνώ με τι ανησυχίε αυτέ. Ε, υπόθηκε ότι είναι προ όφελο των Ευρωπαίων παραγωγών να διασφαλιστεί ένα σωστό μοντέλο για αυτούς. Αυτό όμως απ' την άλλη δεν με έπεισε, διότι θεωρώ ότι θα πληγούν ιδιαιτέρως οι κτηνοτρόφοι παραγωγή βόλου κρέατος αλλά και χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία σε διεθνές επίπεδο. Δεν έχουμε αρκετό προϋπολογισμό και καταβαραθρώνονται οι τιμές και τα εισοδήματα των αγροτών και των παραγωγών. Δεν έχουν πολύ νόημα όλα αυτά και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακούσει πιο προσεκτικά. Ευχαριστώ. Έκθεση Ashworth για την απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή απλουστεύει ε, την γραφειοκρατική επιβάρυνση που υπάρχει σήμερα για τους ε, γεωργούς. Και εγώ θεωρώ ότι μετά από αυτή την έκθεση θα προκύψει μια νέα σχέση ανάμεσα στους ε, φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι κυρίως στα μετακομμουνιστικά κράτη όπως στην Ουγγαρία. Είναι αρμόδιοι λοιπόν για την εφαρμογή της ΑΚΕ και αρμόδιοι επίσης για τις σχέσεις ανάμεσα στους ε, γεωργούς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τρομοκρατήσουμε τους φορείς, πρέπει απλά να συστήσουμε μια νέα σχέση. Και την ευθύνη βέβαια δεν τη φέρουν μόνο οι γεωργοί, αυτοί ε, καλούνται να καταβάλουν ε, τα, ε, τις κυρώσεις, αλλά και το κράτος θα πρέπει να τιμωρείται οποτεδήποτε καθυστερεί να εκταμιεύσει τα κονδύλια στους γεωργούς και οι ε, γεωργοί θα πρέπει να μπορούν να καταφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της ε, έκθεσης Ashworth γιατί πιστεύω ότι αποτελεί απλούστευση και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που έχουν σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Ε, και όλα αυτά είναι απαραίτητα οι Ευρωπαίοι γεωργοί ε, πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τα ωφέλη που προσφέρει η ΚΑΠ, να μην συμβαίνει αυτό που συνήθως συμβαίνει, δηλαδή μια γραφειοκρατική καθυστέρηση. Υπάρχει λοιπόν ε, βούληση να έχουμε απλούστερη διαδικασία, περισσότερο κατανοητή τόσο για τους αρμόδιους φορείς όσο και για τους γεωργούς. Στόχος είναι να καταργηθούν όλες οι περιττές διατάξεις, να υπάρχει μια καλή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις τοπικές αρχές. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, κύριος ε, Πρόεδρε, η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να εξετάζεται συνεχώ κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Γιατί περί τι κανόνε κοστίζουν και σε εμά και στου παραγωγού μα χρόνο και χρήμα. Πράγματα που δεν είναι λογικά και χρήσιμα θα πρέπει να καταργηθούν. Ιδίω αυτό εσύ για την πολύ συχνά πολύπλοκη ε, μέθοδο του cross compliance. Θα πρέπει τα συστήματα να είναι πιο διαφανή η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περνάνε πιο πολύ χρόνο στο χωράφι και όχι στο γραφείο τους. Και ελπίζω η Κομισιόν να κατανοήσει τη σημαντική αυτή είδηση και νόημα της εκθέσης μας. Ευχαριστώ κύριε Τότσο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι πραγματικά είναι δεσμευμένοι με τους παραγωγού της περιφερειάς τους. Ένα από τα κύρια θέματα που ακούμε συνεχώς είναι το θέμα της γραφειοκρατίας που εμπλέκεται στην βιομηχανία αυτή. Κύριο θέμα λοιπόν της νέας ΚΑΠ θα πρέπει να είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Η νομοθεσία θα πρέπει να είναι λογική, κατανοητή για τους παραγωγούς και θα πρέπει να τους περιορίζει από την παραγωγή των τροφίμων. Θα πρέπει να ευθυγραφιστεί η νομοθεσία και να πάρει και ευελιξία για τα κράτη-μέλη. Και πιο σημαντικό είναι να ε, Μιλητούν εδώ η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Το Ελεκτικό Συνέδριο θα πρέπει να δείξει ευελιξία και κοινό νου μάλιστα όταν εφαρμόζει κυρώσεις. Μία δημοσιονομική αναθεώρηση χρειάζεται επίσης για να αξιολογηθεί το κόστος των επιθερήσεων στις παραγωγές και τα χρήματα που καλύπτονται και που ε, ανακτώνται με τις κυρώσεις. Ευχαριστώ κύριε Μακίνη, Σας ευχαριστώ πρόεδρε όταν εισάγαμε αυτό το θέμα της αποπλησίας ε, απλουστευσής λίγοι κατάλαβαν ότι η cross compliance θα ήταν τμήμα της δέσμης που χρειάζεται. Νομίζω είχαμε 17 διαφορετικές οδηγίες εδώ και θα πρέπει να ρωτηθούμε στο σώμα πόσο καλά εμείς νομοθετούμε για την απλούστευση. Υπάρχει ένα συναισθητικό τομέα στον οποίο θέλω να σχολιάσω. Είναι ο τομέα των επιθεωρήσεων. Έχουμε αυτές τις επιθεωρήσεις που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά οι παραγωγοί ε, αντιμετωπίζουν και άλλα επίπεδα ε, ελέγχων από τους, την επεξεργαστική βιομηχανία, από τους μεγαλέμπορους κλπ. Όλα αυτά δεν προσθέτουν όμως αξία ή ασφάλεια στο τελικό προϊόν, ε, αυξάνουμε σημαντικά τη γραφειοκρατία και την ενόχληση των παραγωγών από τους οποίους ε, απαιτείται να συμβάζονται σε αυτού του επιχειρητές. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάκουλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση και πραγματικά έχει έρθει η ώρα ε, για την απλούστευση και την απλοποίηση των διαδικασιών της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτό το καιρό ζούμε ζούγκλα επιδοτήσεων ε, κανονισμών, κανόνων και ο καημένος ο αγρότης στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης δεν καταλαβαίνει καθόλου τι γίνεται και ε, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο για να έχουν εμπιστοσύνη και οι αγρότες μας στην κοινή γεωργική ε, πολιτική και να ξέρουν πού κινούνται και πώς λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή ε, η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένας χυλός. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ οι θολές ε, οι διαδικασίες και τα συστήματα και χρειάζεται οπωσδήποτε απροποίηση. Γι' αυτό λέγω ότι η έκθεση Άσχουρ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτές τις εργασίες. Και η πολιτική να είναι στην υπηρεσία των αγροτών μας. Ευχαριστώ, κύριο κύριος Ευχαριστώ είναι πραγματικά αναζωογονητικό να έχουμε τέτοιες εκθέσεις σαν αυτές που συζητούμε σήμερα που μιλούν για απλοποίηση. Μέχρι τώρα ήταν πολύ περίπλοκη η γεωργική πολιτική. Για όλα τα θέματα χρειάζεται διαπαιδαγώγηση ε, αλλά και απλούστευση των διαδικασιών, όχι περιπλοκή. Μέχρι τώρα περιπλέκουμε τα πράγματα. Όποιος έχει πάει σε συγκέντρωση αγροτών θα γνωρίζει ότι τα έχουν χαμένα από ε, όλες αυτές τις διαδικασίες, τα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώνουν τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους. Και θα πρέπει να πούμε βεβαίω ότι καλυσορίζουμε την έκθεση. Οι αγρότες θα πρέπει να ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία και όχι με τη γραφειοκρατία για να ξέρουμε τι τρόφιμα παράγουν, με ποιο τρόπο και να μπορούμε να τα βρίσκουμε με την ε, ανιχνευσιμότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την απλοποίηση αυτή που προτείνεται. Δεν είναι αυτόματο από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Προχωρούμε στην έκθεση Τρούπελ τώρα. Η κυρία Γιάτε Μάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση Τρούπελ η παράγραφος 34 είναι πολύ σημαντική. Ε, στην τροπολογία 5 όμως έκανα λάθος και δεν ψήφισα όπως θα ήθελα. Ε, ε, θα πρέπει να κοστολογήσουμε και το αποτύπωμα του διοξιδίου του ανθρακά. Και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξανασκεφτούμε την ενιαία έδρα, τη μοναδική έδρα η ε, Βρετανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα το φέρει προς συζήτηση. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν και οι άλλες κυβερνήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, γιατί ε, επιβαρύνεται το περιβάλλον και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μειώσει και το κόστος λειτουργίας τους γιατί περνάμε και κρίση και οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η κυρία Αλφάνο. Mrs. Alfano on the ruler report. Έκθεση Ρούλερ. Ε, Συγγνώμη, ήθελα να κάνω μία εξήγηση ε, για μία άλλη έκθεση και μετά μπορώ να την κάνω τώρα και μετά να δώσω και την επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Ρούλε. Παρακαλώ, προχωρήστε αλλά γρήγορα, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Όσον αφορά την έκθεση της ΣΑΟ, εγώ ψήφισα υπέρ για το θέμα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, γιατί αυτό είναι ε, μέρος των στόχων του 2020. Όλα τα κτίρια που έχουν ενεργειακό ισοζύγιο 0 ε, θα έπρεπε να υποστηρίζονται ε, θερμά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άμεσο μέλλον δεν χρειάζεται να παράγουμε περισσότερη ενέργεια, αλλά να χρησιμοποιούμε καλύτερα την υπάρχουσα ενέργεια. Δεν πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια για να κινηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν άμεσα ε, στην επίτευξη των στόχων τη ενεργειακή απόδοση, χρησιμοποιώντα ε, του οικονομικού πόρου που σήμερα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεγαλύτερη ποσότητα ενέργεια. Όσον αφορά δε ε, τα σχέδια για πυρηνικού σταθμού στην Ιταλία, με κίνδυνο τη δημόσια υγεία, είναι κάτι το οποίο δεν θα το χρειαστούμε αν επενδύσουμε του διαθέσιμου πόρου στην αποδοτική χρήση της ενέργειας. Περνάω τώρα στην εξήγηση ψήφου για την έκθεση Ριούλε. Ε, ψήφισα υπέρ γιατί το Κοινοβούλιο ε, υποστηρίζει την μεγαλύτερη πειθαρχία στις δημόσιες συμβάσεις και για τη δημόσια διοίκηση και για τις επιχειρήσεις, ιδίω τις πιο μικρές που θα διευκολυνθούν στη συμμετοχή τους στις δημόσιες συμβάσεις. Ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι δημόσιες συμβάσεις για να ε, ενισχυθεί η αηφόρος ανάπτυξη μέσω εισαγωγής κριτηρίων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στην προκήρυξη των δημοπρασιών. Ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει ένα σύνολο ε, κανόνων πιο διαφανών και ε, επαρκών για την διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Ο έλεγχος εκ μέρους των πολιτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των δημόσιων πόρων και για την ε, υπεράσπιση των συμφερόντων των συλλογικών φορέων και για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόιτοβα. On Επί της εκθέσεως Ρούλε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 ε, πρόκειται να ε, αντιμετωπίσουμε την διαφθορά και θα πρέπει μάλιστα να είναι ε, αυτό, αυτή η πύλη ανοιχτή και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο έτσι ώστε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ξέρουν τι τιμές προσφέρονται για το κάθε κιλόμετρο αυτοκινητοδρόμου για παράδειγμα κλπ. Επίσης θα θέλουμε να ξέρουμε ποιοι έχουν κερδίσει τους διαγωνισμούς για να μπορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εστιάσουν πάνω τους. Thank you, Madam President. Έκθεση Κέλλερ, η κυρία Μαγκίνες. Και εγώ θέλω να μιλήσω ε, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Από ό,τι λέει ο κανονισμός όμως, αν δεν έχουμε τροπολογίες, δεν μπορούμε να κάνουμε και εξήγηση ψήφου. Μην πάση περιπτώσει. Για την έκθεση Κέλλερ. Βάσει της παραγράφου 44 και 45 και της αιτιολογικής σκέψης Ιώτα Λατινικό, ε, καταψήφισα εγώ την έκθεση, γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ 44. Ε, τι θέλει το Κοινοβούλιο. Πέρσι ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει του γαλακτοπαραγωγού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν σε πολύ δινή θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιγόντω έφερε ε, τις επιδοτήσεις εξαγωγέ εξαγωγές και η μόνη που ε, διαμαρτυρήθηκε ήταν η Νέα Ζηλανδία που δεν είναι και αναπτυσσόμενη χώρα. Γιατί βάλαμε αυτή την παράγραφο στην καλή κατά τα άλλα έκθεση. Δεν εξυπηρετεί ούτε το κοινοβούλιο ούτε του παραγωγού μα, Οι οποίοι αγωνίζονται οι άνθρωποι. Μειώνουμε την παραγωγή στην Ευρώπη και αυτό έχει επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο κύριε Μαγκίνες. Ε, έτσι είναι ο κανονισμός. Ε, η έκθεση αυτή δεν θα έπρεπε να έχει εξηγήσει ψήφου γιατί πράγματα είναι αντροπολογίε. Ε, κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες Είχαμε δυσκολίες με κάποιες από τις προτάσεις αυτές και για το λόγο αυτό δεν ακολουθήσαμε τη γραμμή του ΕΛΚ που θα θέλαμε ε, φυσιολογικά να κάνουμε. Και νομίζω ότι η κυρία ε, εξήγησε τους λόγους ε, τους οποίους συμμερίζομαι. Ελπίζω ότι θα καταλάβει και το ΕΛΚ τη στάση μας αυτή. Αν δεν ψηφίσατε σύμφωνα με τον κατάλογο για την έκθεση ε, Ράνερ, ε, έχουμε πρώτον τον κύριο Μακτάνελ. Βαντάλεν. Ευχαριστώ. Υποστήριξα εγώ την έκθεση αυτή γιατί είναι καλή λύση ε, για τις οδικές μεταφορές. Αυτό που χρειάζεται είναι εναρμόνιση της νομοθεσίας και η ερμηνεία της. Αυτό το βλέπουμε ε, στην παράγραφο 17 όπως τροποποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τους αρμόδιους ε, θεσμούς για την ερμηνεία των άρθρων της νομοθεσίας για να είναι γνωστή και σαφής και να τα ξέρουν αυτά όλοι οι φορείς και όλοι οι μεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα να μιλήσω τώρα για την παράγραφο 27, όπως τροποποιήθηκε. Είναι δυσανάλογη ε, ε, αυτή η ε, ευθύνη που δίνεται στο Eurocontrol Europe θα πρέπει οι οδηγοί να αναπαύονται και να αποδεικνύουν ότι έχουν αναπαυθεί. Ο κύριος Αντωνιώζη τελευταίος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση του που υποστηρίζει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα κενά και σημαντικές παραβιάσεις των κοινωνικών κανόνων για τις οδικές μεταφορές, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Είμαι έτσι υπέρ των μέτρων που προτείνει το κείμενο αυτό ε, Όσον αφορά το θέμα ε, της εναρμόνισης των ε, κυρώσεων για τις παραβάσεις αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα ε, υποστηρίζω το να υπάρχει ένα όργανο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Διακόπτεται τώρα η συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα.